Ο πρόεδρος Λαβία θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Με βάση τους κανονισμούς, επειδή έχουμε κοινή συνεδρίαση, θα αναλάβουμε από κοινού την Προεδρία, το πρώτο μισό ένας και το δεύτερο μισό ο άλλος στις ανακοινώσεις έχουμε διερμηνία σε 21 γλώσσες, μαλτέζικα, ιρλανδικά και Αστανικά δεν υπάρχουν. Έχετε λάβει τα έγγραφα μέσω της εφαρμογής e-meeting και αναμεταδίδεται και ζωντανά η συνεδρίασή μας. Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά, αν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, θα θεωρηθούν ε, τις, τα πρακτικά της 16 Απριλίου και ε, Μαΐου θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα τα πρακτικά της κοινή συνεδρίασης. Σε ό,τι αφορά την ουσία τώρα, θα ήθελα να ζητήσω από τους συγητές, κάποιον από τους συγητές, να κάνουν μια σύντομη εισαγωγή είναι παρούσες οι γήτριες. Θέλουν να μας κάνουν μια σύντομη εισαγωγή για να μας βάλουν στο πνεύμα της ψηφοφορίας. Η κυρία Ζόμερ, η κυρία Μόη. Καλησπέρα, ναι. Αν μπορώ, Παρακαλώ. λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι εγώ και η συνάδελφο Σόμερ μοιραστήκαμε αυτή τη δουλειά και θα ήθελα να πω ότι καταρχάς τα σημεία τα οποία κατήφθηναν αυτές τις σκληρές εργασίες που κάναμε ήταν δύο. Η προστασία και η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών και ε, των ζώων που δεν είναι σε καμία περίπτωση δευτερεύοντα. Η υγεία και η ασφάλεια δεν ε, ε, διακυβεύονται με κανένα τρόπο, το προβλέπουν και οι συνθήκες και εμείς δώσαμε μάχη για να μην υπάρχουν κλωνοποιημένα ζώα και αυτό θα είναι ένας νόμος ο οποίος θα πρέπει να προστατεύει την υγεία των πολιτών και την ευημερία των ζώων. Σας εύχομαι λοιπόν να ψηφίσετε κατά συνείδηση σκεπτόμενοι ότι πρόκειται για ένα νόμο ο οποίος θα προστατεύσει 50 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, 500 συγγνώμη, εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ζόμερ τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μας δίνεται να ευχαριστήσω τη συνεισηγήτρια Τζούλια Μόη, ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας, καθώς επίσης και τους σκιώδεις συζητητές θέλω να ευχαριστήσω από τις δύο επιτροπές για τις πολύ καλές συζητήσεις και ε, τους καλώ όλους και εσά να υποστηρίξουμε τους συμβιβασμούς. Βεβαίω ζητούμε πολύ αυστηρούς κανόνες. Ε, δεν μπορούμε να ανήπτουμε τα σχήρας μας ε, εν ε, αγνία ή αθότητη, επειδή εμείς δεν κάνουμε ε, κλωνοποίηση, υπάρχουν, κυκλοφορούν στην αγορά αυτά τα θέματα και ε, υπάρχουν οι απόγονοι, τα προϊόντα, όποιος είναι κατά της κλωνοποίησης είναι εντελώς κατά. Δεν υπάρχει εδώ λίγον. Οπότε ε, προτείνουμε αυτούς τους συμβιβασμούς στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο έχει αυτό να κάνει με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Βεβαίως είμαστε και υπέρ της ευημερία των ζώων, αλλά είμαστε και υπέρ των καταναλωτών μας που είναι κατά της κλωνοποίησης. Και αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στην εντολή που έχουμε λάβει ε, και στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι όλα αυτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική και τη διοντολογία και μας αφορούν πάρα πολύ. Παρακαλώ λοιπόν να υποστηριχθούν οι συμβαστικές μας τροπολογίες. Σας ευχαριστώ και τις δύο. Τις υπόλοιπες ευχαριστίες μετά το τέλος της ψηφοφορίας. <laughs> Ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Πρώτη συμβαστική τροπολογία. Τις συμβαστικές τροπολογίες τις ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, για την πρώτη συμβαστική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η πρώτη συμβαστική τροπολογία. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 2. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 125. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία της συμβαστικής τροπολογίας 3. Τέλος. Εγκρίνεται η συμβαστική τρία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 21 των εισηγητριών. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 21. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 122. Είναι τρεις πανομοιότυπες τροπολογίες, 22 συγγνώμη, 22 και τις υπόλοιπες που είναι παρόμοιες. Ποιος είναι υπέρ των τριών τροπολογιών, 22, 135 και 136. Τροπολογία 22. Κατά. Κατά. Εγκρίνονται οι τροπολογίες. Τροπολογία 23 των εισηγητριών. Ποιος είναι υπέρ της 23. Κατά. Εγκρίνεται. 151. Ποιος είναι υπέρ της 151 διανατάσσεως της χειρός παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. 151. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική 4. Και περνάμε στην 159. Καταπίπτει. Οπότε πάμε στην 26. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 26. Κατά. Εγκρίνατε. Τροπολογία 20. των συνεισηγητριών. Ποιος είναι υπέρ τη 20. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία 20. 27. Επίσης των συνεισηγητριών. Ποιος είναι υπέρ της 27. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 123. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. «164, 165 και 166 μαζί». Ποιος είναι υπέρ των τριών τροπολογιών. Κατά. Απορρίπτονται οι τρεις τροπολογίες. Τροπολογία 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 167. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 168. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 30. Τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. 14. Τη σύντα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 14 της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 170. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 170. Κατά εγκρίνεται. 171. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 31 των εισηγητριών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 172. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 34 των εισηγητριών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πολύ χαίρομαι γιατί ήρθε η ώρα να δώσω τη σκητάλη της Προεδρίας ε, στον κύριο Λαβία, στον πρόεδρο Λαβία. Ευχαριστώ πολύ. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Κύριε Πρόεδρε, έχασα την κάρτα μου. Μήπως μπορείτε να μετρήσετε και εμένα. Mm. Πέραση της ψηφοφορίας. Έγκρινεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. 70, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 72, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 85. Υπέρ. 85. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αν θέλετε να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93 του κυρίου Ταραμπέλα. Υπέρ. 93. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. τα τρία. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, θέλετε παλήθευση. Ωραία. Επαλήθευση για την ίντα 3. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Λυπάμαι πολύ για σας. Τώρα, οι 95 και 96 είναι ταυτόσιμες, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 4 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 102. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφοφορία για το 3α. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στις εισηγήτριες. No? Dobbiamo sospendere la riunione Emily, e ci vediamo alle 4 con il... Okay. Before closing the meeting... Πριν ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση, θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής ΕΜΒΗ ότι θα ξεκινήσουμε στις 4 με τον Επίτροπο Βέλα. Και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω να είστε εδώ στις 4 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.